η ανάπτυξη, ιδιαίτερα σήμερα εν ώψη των δυσκολιών των οικονομιών που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντι. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό και αύριο στις 12 θα γίνει ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα είναι έκθεση Μίτσελ για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης για αναπτυξιακή συνεργασία, διδάγματα και μελλοντική προοπτική. Η αναπτυξιακή συνεργασία μας είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ δυναμικό. Κάνουμε την περίοδο 7 έως 13 πότε είχαμε μια πρικοδότηση σχεδόν 17 δις για να κατονομήσουμε την ε, φτώχεια και να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας και έτσι να έχουμε δημοκρατική διακυβέρνηση σε τις όμορες χώρες. Στο Κοινοβούλιο παρακολούθησε με προσοχή το πώς λειτουργούν οι επιπτώσεις αυτού του μέσου πολιτικής και χρηματοδότησης σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους. Κατέβασε τώρα τις προτάσεις της για την επόμενη γενιά προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων οι Κομισιόν για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περίοδο μετά το 2013 και τον δίσκο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Οπότε έλαβε ναι, λήφθη αυτή η πρωτοβουλία, ώστε να αναλύσουμε τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από αυτό το όργανο τη Αγία Εργασία, ώστε να μπορούμε να δούμε τι προσδοκίε θα έχουμε για το μέλλον και για το μελλοντικό όργανο, η ΔΕ Αμφισιακή Επιτροπή μα, ομόφωνα είπε ότι χρειάζονται οι εξής αρχές, δηλαδή να έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο το οποίο αποκλειστικά να στοχεύει εις τους στόχους της ε, τη εκρίζωσης τη φτώχεια όπως ορίζει η συνθήκη τη Λισαβόνα και θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις αντισώμενε χώρες. Αυτό το νέο μέσο θα πρέπει βασικά να χρηματοδοτεί κάποια μέτρα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την επί μια αναπτυξιακή αρρωγή και ακριβώ όπω τα έχει θέσει η αντίστοιχη επιτροπή του ΟΣΑ. Η ποσοστό για αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αυστηρότερη από ό,τι προηγουμένω από, από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Όμω δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμεί δεν θέτουμε υπό, υπό αμφισβήτηση τα όσα έχει τάσει ο ΩΣΑ όσον αφορά τη συνεργασία μα με αναδυόμενε αγορέ και κάποιε στρατηγικά αναδυόμενε χώρε. Όμω αυτού του είδου η συνεργασία θα πρέπει να μπει σε κάποιου διάβλου διαφορετικών μέσων πολιτική, ώστε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και να προσπαθούμε να προστατεύσουμε ε, την υφή αυτή, την ιδιομορφία αυτή τη μεξική συνεργασία, παιδεία και, άλλε πολιτικέ θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο. Τουλάχιστον 20% τη χρηματοδότηση για τα σχέδια προγράμματα θα πρέπει να πάνε σε αυτούς τους βασικούς ε, τομείς όπως βασική περίβαση και πολιτική υγείας οπότε θα πρέπει έτσι να έχουμε ε, να εντάξουμε κάποια θέματα όπω το περιβάλλον και με τη διαλλαγή σε όλε τι και για αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε πώ θα έχουμε κάποιο είδου αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα φορολογικά συστήματα και ιδίω για αυτέ τι ανισόμενε χώρε θα πρέπει να δούμε πώ θα υπάρχουν έσοδα με την εσωτερική πολιτική, ούτω να αυτομεθεί έτσι η η φτώχεια και η εξάρτηση. Θα πρέπει μέσα σε αυτό το νέο μεσοπολιτική να χρηματοδοτηθεί όπω πρέπει και έτσι να μπούμε στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αναβαθμισμένο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώ θα πάει αυτό το 0,1% σαν στόχο του, ΕΠ εις αυτό αυτού του στόχου τη αρχή πολιτική, να είμαστε μόνο αποτελεσματικοί, να έχουμε κάποιο συντονισμό καλύτερο μεταξύ κομισιών και κρατών μελών και το Κοινοβούλιο. Επομένω δεν μπορεί παρά να είναι υπέρ του να εκπονηθούν τέτοιες στρατηγικές. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε οικονομίες, δεν, το θέμα δεν είναι να πάμε στα ε, να φτάσουμε σε πρικοδότηση 6 δις ετησίως και δείτε πώς αυτό μπορεί να ωφελήσει από τις όμορες χώρες. Επίσης στις αποφάσεις για το νέο μέσο θα πρέπει, το, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισονομία με το Συμβούλιο Δυνάμει του άρθρου 290 της Λισαβόνας. Θα πρέπει να τηρηθεί αυτό το άρθρο, επομένω θα πρέπει αυτή τη βδομάδα να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο, ούτω ώστε να έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν προσεχώς και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει ευρέως αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης αυτές που εκπονήθηκαν με τρόπο νυφάλιο επί τη βάση της εμπειρίας μας για τις διαπραγματεύσεις που έχουμε ήδη κάνει. 14 κανονισμούς τους κωδικοποίησαμε σε έναν Άρα γι' αυτό και θέλουμε ότι αυτού του είδους η αναπτυξιακή βοήθεια και το σχετικό μέσο πολιτικής θα αποδώσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίτσε, λέει ο Πρόεδρος. Μπασέσκου. Κύριε Πρόεδρε, η εξάλληψη της φτώχειας είναι ένα σημαντικό στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο. Η εφαρμογή κάποιων ε, μέσων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας οδηγεί πιο κοντά στους στόχους της χιλιετίας. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει εξωτερικές αρμοδιότητες για να ολοποιήσει τους στόχους αυτούς, θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες γεωγραφικές και θεματικές θα πρέπει να είναι πιο σαφείς έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε πιο αποτελεσμένοι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες των πολιτών, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αποτελέσουν στόχους χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση κάποιων μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης προτεραιότητα, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ζωής και οι χώρες να εξαρτώνται λιγότερο από την εξωτερική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και για να πετύχουν τους στόχους της χιλιετίας που να την προσπάθειες. Πιστεύω ότι και οι δράσεις που βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές έχουν μεγάλη σημασία. Και χαιρετίζω όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν την αναδάσωση, τη διαφύλαξη των οικολογικών συστημάτων που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων. Το 2006 το Διεθνές Ταμείο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ε, δημιουργήθηκε και ιδιωτικοί πόροι χορηγήθηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες για όλα τα προγράμματα που επιτρέπουν την καταπολέμηση ε, των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και θελήσαμε να εισαγάγουμε αυτό τον μηχανισμό οικολογικής ανάπτυξης που θα επέτρεπε στα κράτη-μέλη να δίνουν πιστώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να ε, το πληρωθήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία κυρία Σαμπόρσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, ο συνάδελφος Μίτσελ είναι ειδικό στα θέματα αυτά από την Επιτροπή ανάπτυξης. Ε, τον γνωρίζουμε και τον συγχαίρω για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Θα ήθελα να μιλήσω ιδιαίτερα για την αρχή της επικουρικότητας. Δεν είναι τα κονδύλια το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε. Η Ένωση επιβάλλει τις δυτικές της αξίες της αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η καλύτερη προοπτική είναι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και όχι μόνο να υποσχόμαστε χρήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλύτερη προοπτική είναι το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν τον πολιτισμό τους και την ίδια ώρα να δώσουμε την δυτική οικονομική βοήθεια στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζαμπόσκα η κυρία Ντάντζιλα και τελειώνει η διαδικασία Καρσδιά για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Όπως είπε και η συγγήτρια, η εκρίζωση της φτώχειας είναι ένας από τους βασικούς στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Χρηματοδότηση που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε μια νέα πρόκληση τώρα για αυτό το μέσο. Δηλαδή, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση της τιμής των τροφίμων που αυξάνεται λόγω της ξηρασίας και λόγω των κερδοσκοπικών επιθέσεων κατά των διεθνών αγορών. Χρειαζόμαστε μια γρήγορη και βέληκτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις απότομες αλλαγές στην αγορά αυτή. Και θα πρέπει να ταιριάξουν τα μέτρα αυτά με του διεθνεί στόχου που έχουν καθοριστεί για το μέσο που συζητούμε. Στα πλαίσια τη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τι προσπάθειε που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε η αναπτυξιακή πολιτική να μπορεί να συνεχιστεί. Και έτσι και ο δημοκρατικό έλεγχο και ο δημοσιονομικό έλεγχο να ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye. Και τέλος θα δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ. Πρόεδρε, καλωσορίζει τα σχόλια του Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτάσει, και με τα χαρά βλέπω ότι συμφωνούμε στα περισσότερα ζητήματα. Πάνω από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τον συνεχή διάλογο που λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου και αυτός ο διάλογος έχει παράγει πολύ καλά αποτελέσματα. Λυπούμεθα μόνο που το Κοινοβούλιο δεν θεωρεί ότι κάποια από τα ψηφίσματά του όσον αφορά το προγραμματισμό ε, έγιναν σεβαστά σε κάθε λεπτομέρεια παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη πλήρω τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όποτε ήταν δυνατόν. Όσον αφορά τη συνεργασία για παγκόσμια δημόσια αγαθά, θα ήθελα να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εν γέννη αυτό ίσω θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές τη, διεθνή για τη βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τέτοια συνεργασία όσον αφορά τα παγκόσμια δημόσια αγαθά στις διάφορες τις αναπτυξιακές. Όμως ένα ε, ξεχωριστό μέσο θα αφορά ε, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνοδεύεται από θεματικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδίκηση. Παρόμοια προγράμμα, παρομοίως προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα πλαίσια ασύλου και μετανάστευσης, από τα θεματικά προγράμματα, θα συνεχιστούν και θα εξακολουθούν να ε, κινούνται προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Δεν πρέπει να αμελούμε ε, τις ε, σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων τομέων. Λοιπόν, το αναπτυξιακό ε, δεν γίνεται όταν ψυχοταμείωνεται θύ εντό του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τι προσπάθειε συζητώντα με τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντα πρωτίστω υπόψη του διάφορου στόχου και αρχέ τη Συμφωνία Κοτονού. Όσον αφορά την χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου Μπαρόσο της 7 η Μαρτίου του 2011 και εδώ ο Πρόεδρος ανέφερε μια νέα αρχιτεκτονική που θα αντικατοπτρίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι η ευελιξία όσον αφορά τη διαδικασία προγραμματισμού, ούτως ώστε η χρηματοδότηση και οι προτεραιότητες όπως αρμόζονται ε, στον κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα σήμερα. Αυτό μπορεί να με την εισαγωγή πολλών κατεξουσότηση πράξεων σεβόμενοι τα κριτήρια που απορρέουν από το άρθρο 290. Εν κατακλείδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελεί χρήσιμη η ζωή συνεισφορά όσον αφορά την ετοιμασία του νέου μέσου στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην εμέσια διάταξη είναι η έκθεση Wallace. Πρόκειται για πολιτικές για τη δέσπιση ενός ευρωπαϊκού